Του ψήφων που έλαβα χώρα σήμερα το απόγευμα. Ε, να σα υπενθυμίσω επίση ότι οι υπόλοιπε επεξηγήσεις ε, ψήφου μπορούν να χορηγηθούν και να κατατεθούν γραπτά. Για την ψήφη για τη σύσταση του κ. Όλμπρεχτ και της κυρίας εαυτό μας για τον κανονισμό του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Είναι Τζίλ η πρώτη. She's absent. Uh... Δεν είναι παρούσα. nařízení rady eh, které upravuje víceletý finanční rámec protože Σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές για την Τσεχία που επιτρέπει γιατί 80 δισεκατομμύρια κορώνες για το 2014 θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και το 2015. Αν δεν συνέβαινε αυτή η αλλαγή στην Τσεχία θα χάνονταν η χρηματοδότηση για το 2014 διότι τότε δεν είχαμε καταφέρει να εγκρίνουμε ούτε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ο κανονισμός εγκρίθηκε αργά. Άλλο πρόβλημα αυτό. Οι αλλαγές λοιπόν που συμφωνήσαμε σήμερα είναι χρήσιμες διότι βοηθούν στην πλήρη χρησιμοποίηση των πόρων για τις φτωχές περιοχές. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Νότης Μαριάς. Υπέρ της τροποποίησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 γιατί έτσι θα μπορούν να μεταφερθούν το 2015 κονδύλια που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν. Θα υλοποιηθούν 300 λειτουργικά προγράμματα. Ειδικότερα σε σχέση με την Ελλάδα θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν προγράμματα για τον περιορισμό της ανεργίας που έχει φτάσει στο 26%. Θα υλοποιηθούν προγράμματα για έργα κοινοφελού εργασία και κατάρτιση χιλιάδων νέων στην Ελλάδα, την ώρα που η ανεργία των νέων μα λόγω τη Τρόικα και των μνημονίων έφτασε στο 51,7% θα χρηματοδοτηθούν επίσης προγράμματα στον πρωτογενή τομέα προκειμένου οι έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος παραγωγής. Μέσα από το Ταμείο Συνοχής θα υλοποιηθούν έργα για υποδομές στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας. Τέλος, η έρευνα, η καινοτομία και η εκπαίδευση θα ενισχυθούν με την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Ε, ε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρώνεται, ολοκληρώνεται η επεξήγηση ψήφου για αυτό το ζήτημα. Τώρα περνάμε στην έκατοντα ετηρίδα της γενοκτονίας των Αρμενίων. Ο κύριος Πόσπισιλ. Ευχαριστώ. Υπερψήφισα διότι το Κοινοβούλιο είναι ένα θεσμικό όργανο που συζητά εκτενώς το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να ε, θυμίσουμε την πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, αυτό το τραγικό γεγονός της ιστορίας ε, του έθνους της Αρμενίας. Θα πρέπει να δημιουργηθεί έτσι μια ευκαιρία για την Τουρκία που παρότι έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε σχέση με το πώς εκλαμβάνει το ρόλο της ε, σε αυτήν την τραγωδία, το πώς προσεγγίζει το θέμα, παρόλο αυτό δεν έχει αναγνωρίσει ότι πρόκειται για γενοκτονία. Χαίρομαι που συμπεριλαμβάνουμε το άρθρο 5 στην, στο ψήφισμα. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ε, ούτως ώστε η Τουρκία να αναγνωρίσει την γενοκτονία σημειώνοντας πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Σκρίπεκ. Ευχαριστώ. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού ε, για την εκατοετηρίδα της γενεκτονίας των Αρμενιών. Η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει δυστυχώς αυτή τη γενοκτονία στην οποία χάσαν τη ζωή τους 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Η γενοκτονία θα πρέπει να αναγνωριστεί προκειμένου η Τουρκία να μπει στον δρόμο της συμφιλίωσης και στον δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τελική ανήλυση να μπορέσει να προχωρήσει. Η Τουρκία θα πρέπει να κατανοήσει στην τελική ανάλυση ότι είναι χρήσιμη η μεταμέλεια και η αντιμετώπιση του παρελθόντος. Θα πρέπει να το κατανοήσει λοιπόν και ότι η άρνηση της πραγματικότητας ε, ουσιαστικά αποτελεί διάγνωση για την επανάληψη των σφαλμάτων στο μέλλον. Για να μην επιτραπεί στο μέλλον ποτέ ξανά τέτοια εγκλήματα. Ε, νένι δαμα Μιχαήλα Σόιντροβα. Κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστήριξα το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων που εκφράζει και την ανάγκη ωστόσο συμφιλίωσης μεταξύ Αρμενίων και Τούρκων. Δεν είμαστε δικαστήριο όμως. Είμαστε υποχρεωμένοι να δείξουμε την άποψή μας σε τέτοια σημαντικά γεγονότα χώρες και τα κατεστημένα των χωρών που το έκαναν πρέπει να το κάνουν. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και το αδίκημα και να παράσχουμε συγχώρηση. Το κάνανε οι Γερμανοί, το κάνανε άλλοι. Εμείς ζούμε την 70η ε, επέτειο ενός από τα μεγαλύτερα αδικήματα, ενός, ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ιστορία των γερμανο-τσεχικών σχέσεων. Ξέραμε πόσο χρειάστηκε να ε, παλέψουμε γι' αυτό. Θα ήθελα η Ερμενία και η Τουρκία να τα βρουν. Ο κύριος Μίκα έχει το λόγο. Με μικρόφωνο. Με μικρόφωνο. Συγγνώμη. Εμείς απόσχομεν, διότι δεν ξέρουμε πώς να ψηφίσουμε. Στην Πολωνία δεν υπάρχουν αισθήματα κατά τον Ρωμά, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι... Ε, συγγνώμη, κοιτάξτε, ε, ε, δεν μιλούμε για τους Ρωμά, αλλά για την Αρμενία. Άλλο οι, Αρ, Αρμένοι, άλλο οι Ρωμά. Είστε, έχετε ζητήσει να κάνετε εξήγηση ψήφου, αλλά μιλάτε για τους Ρωμά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Περιμένετε το επόμενο θέμα να μιλήσετε όταν γίνει η συζήτηση για τους Ρωμά. Ο κύριος Μαριάς. Υπερψήφισα το ψήφισμα με το οποίο αναγνωρίζεται η γενοκτονία των Αρμενίων γιατί έτσι μπορούμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στα εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά των Αρμενίων που σφαγιάστηκαν από τα στρατεύματα των Νεότουρκων που στόχο είχαν την εθνοκάθαρση. Εκατό χρόνια μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων η ανθρωπότητα κλείνει το γόνι στον τάφο του, Από του απλού πολίτε του κόσμου μέχρι τον Πάπα όλοι με ένα στόμα καταδικάζουν τις μαζικές σφαγές των Αρμενίων, καταδικάζουν αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητα. Η υπερψήφιση λοιπόν του ψηφίσματος συνιστά όχι μόνο μια αποκατάσταση της αλήθειας, αλλά μια ιστορική πράξη που ασκεί πίεση στην Τουρκία, που πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, αλλά και την γενοκτονία των Ποντίων και να ζητήσει συγγνώμη. Οφείλει να δεσμευτεί στην πράξη η Τουρκία ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο αποσύροντας τα τουρκικά στρατέματα κατοχής από την Κύπρο και έροντας το κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας. Ευχαριστώ. Η άρνηση της γενικονίας των Αρμενίων είναι σε κάποιες περιπτώσεις ποινικά διώξιμη και αυτό το υπόδειγμα θα πρέπει να το, το παράδειγμα θα πρέπει να το ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Μόνο αναγνωρίζοντας την γενεκτονία μπορούμε να διδαχτούμε από τα φρικτά εγκλήματα του παρελθόντος. Γιατί αρνούμενοι το κακό είναι σαν να αφήνουμε μια πληγή να ματώνει. Στην ψηφοφορία λοιπόν ψήφισα υπέρ των ε, τροπολογιών εκείνων που μας υπενθυμίζουν τα ευθεία αυτά λόγια. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να ιαθούν οι πληγές του παρελθόντος. Ε, ε, Ο κύριος Τίμπορ Ευχαριστώ. Υπερψήφισα το ψήφισμα διότι θα μας θυμίσει ξανά το πού μπορεί να οδηγήσει ο υπερβολικός εθνικισμός. Είναι ανησυχητικό το ότι εμφανίζονται ρητορικές, ακροδεξιές, ε, εναντίον των μειονοτήτων, των Ρωμά, ανά την Ευρώπη. Συχνά αυτές οι θέσεις γίνονται εγκτές και υποστηρίζονται από ηγέτες και κυβερνήσεις. Θα είχα προτιμήσει να υπάρχει εντονότερη η αναφορά στον κίνδυνο του εθνικισμού. Ωστόσο με το κείμενο αυτό ε, νομίζω η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει ένα σαφές μήνυμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όμπερ Μαρία. Στην ε, Βιέννη Πρόταρτε για την ε, πρώτη παρουσίαση σε λογοτέχνημα της γενοκτονίας των Αρμενίων. Σήμερα όμως, τόσο χρόνια μετά, η Τουρκία ακόμα αρνείται με ρητορικές. Ο Παπας Φραγκίσκος μίλησε με λόγια και αυτό που μου φαίνεται πολύ ε, αμφιλεγόμενο είναι ότι όχι μόνο οι Ισλαμιστές άρνουν την ιστορία της αλλά ακόμα και η τουρκική νεολαία στην Ευρώπη κατηγορεί όλους όσους ε, υποστηρίζουν την γενεκτόνια των Αρμενίων. Είναι πολύ απλητικό αυτό ότι ακόμα και στην τρίτη γενιά δεν έχουν καταφτάσει ακόμα στην δημοκρατική Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν ε, και υποστήριξα σήμερα το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ταμπάσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα για πολλούς λόγους. Ε, πρώτα απ' όλα, συμπάσχω ε, για τις οικογένειες αυτών των εκατομμυρίων Αρμενίων ε, που ήταν τα θύματα της γενοκτονίας. Μην ξεχνάτε ότι στην Οθωμανική μετά τη πτήρωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τους ε, νεότουρκους έπεσαν θύματα αυτής της γενοκτονίας όταν οι νεότερκοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια νέα εθνική ταυτότητα. Τώρα λοιπόν θα πρέπει πολιτικός πώς και οικονομικός να επομιστεί η Τουρκία την ευθύνη της και να αποζημιώσει τους ε, ε, το... τα θύματα των γενοκτονιών που ε, προέρχονται από διάφορα έθνη, από την Αρμενία, από τη Βουλγαρία, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια ποινική δίωξη, κυρίως να μην αρνείται η ύπαρξη ε, αυτού του γεγονότος. Σας ευχαριστούμε. Τώρα θα ακολουθήσουν ε, οι επεξηγήσεις ε, ψήφου για το ψήφισμα της Διεθνούς ημέρας για τους Ρωμά και για τη γενοκτονία των Ρωμά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πρώτος ομιλητής μας είναι ο Μπράνισλαφ Σκρίπεκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού για τη γενοκτονία των Ρωμά δεν θα πρέπει να ξεχαστεί όπως κάθε άλλη γενοκτονία όχι μόνο ως υπενθύμηση των φρικαλαιοτήτων αλλά και ως κίνητρο να ταχθούμε υπέρ της κοινότητας αυτής. Η κοινότητα το Ρώμα και η εκπροσωπή της και στη Σλοβακία έχουμε πάνω από 400.000 Ρωμά. Καθημερινά είμαστε αντιμέτωποι με το θέμα της ένταξης των Ρωμά. Και βασική αιτία της ε, αποτυχίας της ένταξης είναι και η κοινότητα των Ρωμά. Θα πρέπει να συμμετέχουν πιο πολύ οι Ρωμά και θα πρέπει να συμμετέχουν και στην πολιτική και στην εκπαίδευση. Γιατί η άσκοπα χαλάμε τα λεφτά μας. Το 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε μια ιστορική απόφαση. Αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ρωμά που δολοφονήθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς και τους συνεργάτες του, μια και θεωρούσαν τους απανταχού Ρωμά ως φυλετικά κατώτερους συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από τότε που οι Ρωμά κατά χιλιάδες σύρθηκαν στα κρεματόρια των ναζιστικών στρατοπέδων, στο Auschwitz, στο Νταχάου, στο Μπέλσεν, στο Μάουτχάουζεν, εκεί όπου δολοφονήθηκαν και χιλιάδες Έλληνες πατριώτες. Υπερψήφισα λοιπόν το ψήφισμα που καταδικάζει την γενοκτονία των Ρωμά από τους Ναζί, γιατί θεωρώ ότι έτσι τιμούμε τη μνήμη χιλιάδων Ρωμά που δολοφονήθηκαν μαζικά από τους Ναζί, στέλνοντας ταυτόχρονα αποφασιστικό μήνυμα στους κάθε λογής νοσταλγούς του ναζισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Μαριά. Τελευταίος, αλλά εξίσου σημαντικός, ο κύριος Κόρβιν Μίκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πήγα ε, ότι δεν ήξερα πώς να ψηφίσω, διότι δεν υπάρχουν τέτοια ε, προβλήματα στην Πολωνία. Ακούμε τους τσιγκάνους να τραγουδούν, να χορεύουν, να παίζουν ε, βιολιά. Ε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι με τους Ρωμά που ε, απομιζούν τα λεφτά από το σύστημα εθνική εθνικής ασφάλισης που μένουν σε ε, άθλια διαμερίσματα. Το θέμα είναι ότι άλλο η Ρώμα, άλλο οι Τσιγκάνοι, οι Αθήγανοι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα τσακωθούμε τώρα για αυτό το θέμα. Ήσασταν είναι και ο τελευταίο ομιλητής στις επεξηγήσεις ψήφου. Καιρό είναι να κλείσουμε την συνεδρίαση. Τα πρακτικά